Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλώς ορίσατε αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ να καθίσετε. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. της Ρέτζη για σήμερα, 9η Νοεμβρίου. Υιοθέτηση της ημερήσιας διάταξης. Εδώ έχω μία παρατήρηση να κάνω για την πρόταση που έχετε μπροστά σας. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι μου ζήτησε η ψηφοφορία για την έκθεση πρωτοβουλίας του για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 16 να γίνει η ψηφοφορία στην επόμενη συνεδρίασή μας στις 29 Νοεμβρίου. Εγώ δέχθηκα το αίτημα αυτό. γιατί νομίζω ότι με αυτές τις εκθέσεις θα πρέπει να είμαστε επακριβείς και αν απαιτείται περισσότερος χρόνος γιατί όχι. Το τμήμα αυτό των ψηφοφοριών λοιπόν διαγράφεται, αναβάλλεται μάλλον, μέχρι τη συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου. Με αυτή την αλλαγή παρακαλώ να δεχθείτε την ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Μποστινάρο. Α, όχι, τη δέχεστε. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Έχουμε την ημερήσια διάταξη για την σημερινή και την αυριανή συνεδρίαση. Έγκριση των πρακτικών τώρα, της 8 η Σεπτεμβρίου και της 11 ε, ε, η Οκτωβρίου. Η πρόταση για τα πρακτικά είναι, ε, είναι διαθέσιμη online. Αν δεν υπάρξουν αντιρρήσει κατά τη διάρκεια της ε, συνεδριάσεω αυτής ε, θα, γίνουν δεκτά, θα θεωρηθούν δεκτά άμα το τέλος της. Λοιπόν, περνάμε τώρα στι ανακοινώσει του Προέδρου. Έχω μία ανακοίνωση να κάνω και νομίζω ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον για σας. Αφορά στη συνεδρίαση Habitat 3 στο Κίτο. Δύο από τα μέλη μας είναι στην αντιπροσωπεία την οποία δημιούργησε η Επιτροπή ΤΕΒΕ, Όλμπριχτ και Βέστφαλα. Θα τους δώσω το λόγο να μας κάνουν μια μικρή ενημέρωση. Να ξεκινήσω με τον κύριο Ολμπριχτ. Γιατί έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις αμέσως μετά. Έχετε το λόγο κύριε Ολμπριχτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα δώσω κάποιες γενικές πληροφορίες και η Βέσφαλ θα σας δώσει τις λεπτομέρειες, μιας και είναι εισηγήτρια για τα θέματα Urban. Η συνάντηση Habitat 3 λοιπόν οργανώνεται από το Habitat Ηνωμένων Εθνών κάθε 20 χρόνια ήταν μια έκτακτη συνεδρίαση, δεν είναι κάτι το συνηθισμένο. Και οι στόχοι αλλάζουν και η ατμόσφαιρα γενικά αλλάζει. Αυτό το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον στην παρούσα φάση είναι ότι βασίζεται πλέον στους στόχους της αηφορίας των Ηνωμένων Εθνών. Έχει σημασία αυτό ιδιαίτερα για τον στόχο 11. Και στα πλαίσια του στόχου 11 για την αηφορία η ομάδα Ηνωμένων Εθνών για το Habitat έχει ε, θέσει το θέμα της εξέτασης της αστικοποίησης ε, στον κόσμο και γενικά η συζήτηση για τις αστικές περιοχές, οι αστικοποιημένες περιοχές. Ε, τέθηκε το θέμα στο Κίτο λοιπόν. Αυτό το οποίο πολιτικά έχει στην παρούσα φάση ενδιαφέρον είναι ότι η προσπάθεια αυτή γίνεται εδώ και μήνες έτσι ώστε να πισθούν τα Ηνωμένα Έθνη ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στοιχεία όχι μόνο για τους πολίτες, τους ίδιους, αλλά και τη διακυβέρνηση των αστικών περιοχών. Γιατί? Γιατί η τοπική δημοκρατία και οι τοπικοί άρχοντες και αρχές αντιμετωπίζονται από τις δομές των Ηνωμένων Εθνών σαν μικιό. Γι' αυτό ακριβώς και η συζήτηση που γίνεται γύρω από τις τοπικές αρχές αφορούσε περισσότερο στις ΜΚΙΟ, δεν είχε καμία σχέση με τους τοπικούς άρχοντες. Για αρκετούς μήνες λοιπόν γινόντουσαν συνεχείς προσπάθειες από πάρα πολλές ε, οργανώσεις ε, τοπικών αρχών, ιδιαίτερα το Παγκόσμιο Δίκτυο, το οποίο έχει δημιουργηθεί και, από, και συναποτελείται και από ευρωπαϊκά δίκτυα, έτσι ώστε να πισθούν τα Ηνωμένα Εθνή να συζητηθούν τα θέματα της ανάπτυξης των αστικών περιοχών. Ευφυής πόλεις, σαν παράδειγμα. Από την άλλη, πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα της διακυβέρνησης των περιοχών αυτών. Γιατί αν δεν μιλήσουμε για τη διακυβέρνησή τους, τότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε λοιπόν στο Κίτο ήταν ότι η συζήτηση διεξάγεται σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο αφορά τα θέματα γύρω από τις πόλεις, ε, μεταφορές, εφής, πόλεις, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και το δεύτερο επίπεδο είναι το λεγόμενο δικαίωμα της πόλης, ή δικαιώματα των πολιτών, των επιχειρήσεων κτλ. Το ένα επίπεδο είναι λοιπόν το τι θα κάνουμε με τις αστικές περιοχές και το άλλο επίπεδο είναι η διακυβέρνηση των αστικών περιοχών. Ήταν ενδιαφέρον ότι οι Ευρωπαίοι, αλλά σαν παράδειγμα και οι Συγκαπούροι και άλλοι, ασχολήθηκαν με τις εταιρικές σχέσεις, την ενιαία αντιμετώπιση, ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Από την Αφρική αναφέρονται στην ανάγκη για την αποκέντρωση σαν παράδειγμα, γιατί δεν υπάρχει καμία τάση αποκέντρωσης. Συνεπώς λοιπόν για τις χώρες αυτές η επίλυση των προγραμμάτων αυτών, των προβλημάτων των αστικών περιοχών, σημαίνει ότι θα ενισχυθεί η τοπική δημοκρατία και οι τοπικές αρχές. Είναι σαφές λοιπόν ότι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν πολύ καλά στο Κίτο, μιλούσαν σε ένα λίγο διαφορετικό επίπεδο. Εμείς μιλούσαμε για τον κίνδυνο εκ νέου συγκεντρωτική αντίληψης, ενώ αυτοί είχαν τον αρχικό στόχο της αποκέντρωσης. Από κοινού όμως τέθηκε η προβληματική των αστικών περιοχών. Και μια τελευταία παρατήρηση από πλευράς μου. Ίσως ήταν ένα καλό βήμα που υπήρχε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι του Κοινοβουλίου, όχι της Επιτροπής, αλλά της Ένωσης. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων είχαμε επίσης και τα εγγένεια μιας ευρωπαϊκής έκθεσης, η οποία ήταν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι της Ένωσης. Είπαμε λοιπόν στους συναδέλφους ότι την επόμενη φορά θα πρέπει να είναι έκθεση της Ένωσης και όχι μόνο της Επιτροπής γιατί αν μιλάμε μόνο για την Επιτροπή, τότε θα έπρεπε να έχουμε ένα διαφορετικό στάντ εμεί. Εν πάση περιπτώσει αυτά έγιναν. Νομίζω ότι η συνδυασμένη αντιμετώπιση, η αποκοινού αντιμετώπιση είναι ένα πολύ καλό βήμα. Λοιπόν, κλείνοντα τη δική μου αντίδραση, τη δική μου παρέμβαση, η Ευρώπη εκπροσωπήθηκε σωστά. Η Ευρώπη παρουσίασε πράγματι κάποια, κάποιες θετικές κατευθύνσεις και αποδείξαμε ότι ήδη έχουμε κάνει πολλά στην Ευρώπη στον συγκεκριμένο τομέα. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να αποφασίσουμε και να αποφύγουμε είναι το εξής. Δεν θα πρέπει σε αυτές τις συνεδριάδες να λέμε ότι θα πρέπει να μας ακολουθήσετε, γιατί αν το κάνουμε αυτό χάσαμε. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι πρέπει να συνεργαστούμε μαζί σας και να συμμεριστούμε τις εμπειρίες μας γιατί αλλιώ όταν λέμε θα πρέπει να κάνετε ό,τι εμεί μα κατηγορούν για νέο απεικιοκράτε και η συζήτηση έχει λήξει. Λοιπόν, πρέπει να του δείξουμε ότι πολλέ φορέ μαθαίνουμε και από αυτού, γιατί έχουν νέε ιδέε, σύγχρονε ιδέε, είναι πολλοί επαγγελματίες, ικανότατοι, νομικοί σαν παράδειγμα από την Αφρική. Έχουμε πολλά να μάθουμε και από αυτού. Σα ευχαριστώ. Κυρία Βέστφαλ.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 όχι μόνο ως Ευρωπαίοι, αλλά και η παγκόσμια κοινότητα γνωρίζει πως τα ερχόμενα χρόνια τρία τέταρτα του πληθυσμού στις πόλεις θα ζουν στις πόλεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε μικρές, μέσες και μεγάλες πόλεις, αλλά και σε μεγαλοπόλεις λεγόμενες megacities. Γι' αυτό και οι εκδηλώσεις τη UN Habitat δεν πρέπει να γίνονται ανά 20 χρόνια, αλλά ανά συντομότερα χρονικά διαστήματα, το οποίο και έγινε. Επειδή αν δεν γινόταν αυτό, δεν θα, ήταν παρά, δεν θα είχαμε παρά μια επιφανειακή ενασχόληση με το θέμα. Δεν είναι μόνο το γεγονός πως το ατρέταρτα του πληθυσμού Εκεί θα γίνουν πολλά. Ένα επίκεντρο είναι παραδείγματος χάρη επίσης η πολιτική που απευθύνεται στα παιδιά. Μπορείτε να συγχωρέσετε με, αλλά σήμερα όταν ξύπνησα ένιωσα ένα χτύπημα στο πρόσωπο. Επίσης ήταν μια σφαλιάρα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδίω αν σκεφτεί κανεί τη νέα πολιτική για τα παιδιά που θα ασκηθεί στι στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή ο κύριος Τραμπ ως νέος πρόεδρος προανήγγειλε πως δεν αισθάνεται υποχρεωμένος απέναντι στα παιδιά, αλλά αυτό ήταν ένα σημαντικό ζήτημα που έπαιξε ρόλο στο Κίτο. Επειδή είναι αυτονόητο πως στις πόλεις η κλιματική πολιτική πραγματοποιείται σε διάφορα επίπεδα. Γι' αυτό και αυτό που ανέφερε και ο Γιάνν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκπροσωπείται όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό και θα είχε ζήτημα να το κάνουμε από κοινού ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή ως Ευρωπαίοι και με αυτό που αποφασίσαμε ως ατζέντα πόλεων, Πρέπει να ελέγξουμε λοιπόν ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Επειδή δεν είχαμε μόνο θετικό feedback για το μοντέλο, αλλά υπήρξαν και περιπτώσεις που αναγκάσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αλλάξει πράγματα και να δραστηριοποιηθεί για εταιρικές σχέσεις και για μοντέλα εταιρικών σχέσεων και γι' αυτό άκουσαμε θετικά λόγια και πιστεύω πως βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο και αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε και εκεί έχει δίκιο ο Γιάν, είναι να δείχνουμε με το δάχτυλο και να κάνουμε τους ξερόλες. Δεν είμαστε ξερόλες, δεν τα ξέρουμε όλα, αλλά μπορούμε να κάνουμε προτάσεις, μπορούμε να συμμετήσουμε δίκτυα και μπορούμε να παρουσιάσουμε σε άλλους πράγματα που λειτουργούν καλά σε εμάς. Τώρα το αν θα το αποδεχτούν αυτό απόκειται στις πόλεις τις ίδιες. Ευχαριστώ πολύ. Yeah, of Μόλις τέλειωσε η συνεδρίαση με την έγκριση της νέας ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τις αστικές περιοχές και είναι καλό οι συνάδελφοι να έχουν το κείμενο αν το αναζητήσουν. Στο έγγραφο αυτό λέγεται ότι τα μέτρα τα ευρωπαϊκά τα οποία έχουμε ήδη προτείνει είναι η βάση και για το ευρύτερο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι τυχαία η συμπληρωματικότητα. Σαν παράδειγμα το θέμα των εφιών αστικών περιοχών είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και για τα Ηνωμένα Έθνη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση που τα πρώτη είναι πρώτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν την τελευταία μέρα παρουσίασαν και τις υποχρεώσεις τις οποίες θα πρέπει να αναλάβουμε για να πετύχουμε τους στόχους στα πλαίσια ε, της χιλιετίας, των στόχων της χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι η νέα ατζέντα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περάσει και από την αντίστοιχη των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκαθαρίζει τις θέσεις της και ενισχύει τη συνεργασία ανάμεσα στις πόλεις στον τομέα της αηφορίας. Λοιπόν, αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό, γιατί είναι σημαντικό και για τον κόσμο, αλλά είναι πολύ σημαντικό και για αυτά τα οποία έχει ήδη κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλάμε για τις ανηλυμένες υποχρεώσεις εισαγωγικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γύρω από αυτό. Ευχαριστώ, συγχαρητήρια λοιπόν στους δύο εκπροσώπους μας στο Κίτο για το Χάμπιτα 3. Είμαι σίγουρη ότι πράγματι εκπροσωπήθηκε περίφημα η Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό. Θα παρακολουθήσουμε τη διαδικασία προσεκτικά και για την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών και για την αντίστοιχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποια σχόλια. Τότε περνάμε στις ψηφοφορίες, παρακαλώ. Όπως είπαμε, αναβλήθηκε το ένα τμήμα των ψηφοφοριών και γι' αυτό θα ψηφίσουμε σήμερα την έκθεση του κυρίου Τσίκου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Αξιολόγηση. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μια έκθεση για την εφαρμογή τον προηγούμενο χρόνο του Ταμείου. Τον Οκτώβριο του 2015 δημοσιεύθηκε η νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειτουργία του Ταμείου το 2014. Χρησιμοποιήσαμε την ευκαιρία αυτή για να συντάξουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας αξιολογώντας τη μέχρι τώρα λειτουργία του Ταμείου. Μετά από τις παρουσιάσεις αυτές, η Επιτροπή δημοσίευσε τη δική της έκθεση το 2015. Ο εισηγητής μας έλαβε υπόψη την έκθεση λοιπόν του 2015 και ε, συμπεριέλαβε και τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Έχουμε γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής ε, Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου. Έχουμε και 15 συμβιβαστικές οι οποίες συνετάχθηκαν σε συνεργασία με τους Σκιώδης. Κύριε Τσίκου, δέλετε το λόγο. έχετε το λόγο, Τσίκου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι πράγματι νομίζω ότι κάναμε καλή δουλειά. Πράγματι προσπαθήσαμε να εντάξουμε με ισόρροπο τρόπο και με αντικειμενικότητα όλες ε, τις πλευρές οι οποίες κατ' εμέ είναι κομβικές για την ανάγκη μείωσης του χρόνου παρέμβασης και Προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε λίγο την φύση των παρεμβάσεων ανάλογα με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν ε, κατηγορίες του πληθυσμού και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί που διαχειρίζονται τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ ε, όλους για την προσφορά τους και την συνεργασία τους. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες τώρα. Θα ξεκινήσουμε με τη συμβιβαστική 4. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές γίνεται δεκτή. Περνάμε τώρα στη 34. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 38. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, Δεκτή. 51. Υπέρ. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Για, συγγνώμη. Το πρώτο τμήμα της 51 επαναλαμβάνει η πρόεδρος, επαναλαμβάνει την ψηφοφορία για το πρώτο τμήμα της 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ α, όχι, το δεύτερο τμήμα δεν ψηφίζεται. Θα περάσουμε τώρα στη συμβιβαστική 9, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Συνεχίζουμε με την 57. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συνεχίζουμε με την 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές δεκτή 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συγγνώμη, συγγνώμη. Δεκτή. Η 70 γίνεται δεκτή. 70 γίνεται δεκτή. 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 98. 98. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 100. Προφορική τροπολογία. Έχετε κάποια αντίρρηση για την προφορική τροπολογία. Όχι. Συνεπώς ψηφίζουμε. Την 100 συμπροφορική προφορική υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 108. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 109. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τρία υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Συγγνώμη. Την τροπολογία αυτή την υποστηρίζει ο εισήγητης. Εν πάση περιπτώσει, ηλεκτρονική κλίση για την τροπολογία υπαρίθουν τρία... Ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. Δεκαοκτώ κατά δεκαεπτά υπέρ. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 5 υπέρ κατά αποχές απερίφη. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. δεκατρία υπέρ κατά αποχές απερίφη. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε τώρα στη συνέχεια στις προτάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Η... Ξεκινάμε λοιπόν, η A και η B καταπίπτουν, C υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. D υπέρ, κατά, αποχές απερίφθη ή υπέρ κατά αποχές απερίφθη Εφ υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική κλίση 4 Ψηφίζεται. Πέρας. Απερίφθη. Πέντε. Υπέρ. Πέντε. Επαναλαμβάνω. Ε, κατά. Αποχές. Απερίφθη. Τώρα περνάμε στις προτάσεις της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών. Ένα. Υπέρ. Κατά. Ε, α, έχει καταπίσει η αιτιολογική σκέψη ένα. Η D, αγγλικό D, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ή, e, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Ένα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Δύο Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Η τρία, Σε δύο τμήματα το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Περνάμε τώρα στην 7. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Η 8. Υπέρ, κατά, αποχές, απερίφθη. Η 9. Η υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 12. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 13 σε δύο τμήματα. Το δεύτερο ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απερίφη Και η 15. Υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τώρα περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορίες. Γίνεται δεκτή λοιπόν. Συγχαρητήρια στον κύριο Τσίκου. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Okay, we can continue. Ευχαριστώ. Μπορούμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα σημεία της ημέρησιας διάταξης. Επόμενο θέμα είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Ενρίκο Ρώση, αντιπρόεδρο, και τον Νίκολας Μπρούξ, διευθυντή για την πολιτική συνοχή της διάσκεψης των παράκτιων περιφερειακών περιοχών της Ευρώπης. Η διάσκεψη αυτή θεσπίστηκε το 1973. Πρόκειται για μια ομάδα προβληματισμού και άσκηση πιέσεων για τι θάλασσες περιοχές. 160 περιοχές εκπροσωπούνται από 28 χώρες και μέλη της Ένωσης και μη μέλη της Ένωσης. Έχουμε και έξι γεωγραφικές περιοχές, η CBMR, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της οργανωτική δομή και προωθεί οργανωτικά προγράμματα μεταξύ των μελών της περιοχής και συζητά θέματα καινού ενδιαφέροντος. Σήμερα θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων για το έργο της διάσκεψης με τους δύο κυρίους που προανέφερα, στους οποίους και θα δώσω το λόγο. Έκαστος θα κάνει μία σύντομη δήλωση, 10 λεπτών καθένας και μετά θα έχουμε ως βουλευτές τη δυνατότητα να υποβάλουμε τις ερωτήσεις μας στους δύο κυρίους. Ο κύριος Ρώση έχει καταρχάς το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιόλογα μέλη της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας εξ ονόματος της διάσκεψης θαλασσίων και περιφερειακών περιοχών θα ήθελα και εγώ να βοηθήσω τις εργασίες σας. Η CRPM, της οποίας είμαι αντιπρόεδρος, είναι μια πολιτική οργάνωση που αντιπροσωπεύει 150 περιοχές στην Ευρώπη. Πιστεύουμε ιδιαίτερα στην πολιτική συνοχή. Θέλουμε να είναι λειτουργική, θέλουμε να την ανανεώσουμε και θέλουμε να υπενθυμίσουμε και όλα τα θετικά τα οποία προκαλεί και που βασίζονται σε τρεις βασικές αρχές, την αλληλεγγύη, την εδαφικότητα και την κοινωνικο-οικονομική ολοκλήρωση. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Γενική μας Συνέλευση υιοθετήσαμε ένα πρώτο έγγραφο για το τι θα ακολουθήσει μετά το 2020. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα, ρίξω ένα βλέμμα στο παρελθόν. Η πολιτική συνοχή δημιουργήθηκε έτσι ώστε όλες τι περιφέρειες της Ευρώπης να είναι σε θέση να πάρουν μέρο στην ενιαία αγορά. Στόχος είναι η αντιστάθμιση ε, των ανισοτήτων και των στρεβλώσεων που μπορούσαν να δημιουργηθούν, βρώντας σε επίπεδο ανάπτυξης περιφερειακό. Η ενιαία αγορά είχε απαιτήσει, αν θέλετε, για να μπορέσει να λειτουργήσει καλά, μια πολιτική συνοχή και επανεξισορρόπηση. Σήμερα η χρηματοπιστωτική κρίση, η οικονομική κρίση και η κοινωνική κρίση απαιτούν περισσότερη πολιτική συνοχή. Για να ελαφρυνθούν οι επιπτώσεις της κρίσης στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης και στις πιο φτωχές αλλά και στις προχωρημένες οικονομικά. Θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε ότι η πολιτική συνοχή είναι η μοναδική πολιτική δημόσια επενδύσεων που αφορά σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Γνωρίζουμε και το λέει η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι κάθε ευρώ επενδύσεων στην περίοδο 2007-2013 είναι ικανό να μοχλεύσει 3 ευρώ επιπλέον ΑΕΠ μέχρι το 2020. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη είναι πλέον προτεραιότητα. Η έννοια αυτή της ανάπτυξης την υπενθύμησε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης δεν υπήρξε καμία συγκεκριμένη αναφορά στις πολιτικές συνοχής και στα διαφορετικά ταμεία. Ας ελπίσουμε ότι ήταν μια απλή αμέλεια. Πάντως καλό θα είναι να γνωρίζουμε όλοι ότι οι περιφέρειες εργάζονται και προσπαθούν όσο μπορούν καλύτερα για να δαπανίσουν σωστά τις πιστώσεις και να πετύχουν τους στόχους τους. Και η δική μου περιφέρεια, η Τοσκάνη, όπως και πολλές άλλες, έχουν ήδη προκαταλάβει αν θέλετε την παρέμβαση των πολιτικών συνοχής έτσι ώστε να γίνουν δεκτές οι προτάσεις προγραμμάτων τους από πλευράς των κοινοτικών οργάνων. Για να είμαστε έτοιμοι δηλαδή όταν τα χρήματα φτάσουν στα ταμεία του κράτους και των περιφερειών. Έχουμε κάνει πρόβλεψη δηλαδή για αυτές τις εισφορές να μου επιτρέψετε να έχω και κάποιες επιφυλάξεις για την πρόταση την οποία ακούμε και που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 επιτρέποντας στις διάφορες χώρες και περιοχές την δυνατότητα να χρησιμοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις αυτές και για διαφορετικούς λόγους από αυτούς οι οποίοι συμφωνήθηκαν θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα αν πράγματι θέλουμε να ασκήσουμε διαφορετικές πολιτικές που απαιτούν άμεση παρέμβαση όπως τον τομέα της μετανάστευσης ή και άλλα θέματα κατεπήγοντα κοινωνικού τύπου αν είναι επαρκές το 1% του ΑΕΠ. Είναι μια πρόταση για σκέψη ε, γιατί εδώ και χρόνια δεν γίνονται βήματα προς τα εμπρός στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Ίσως ε, να έχουμε κάνει βήματα προς τα πίσω και αυτό αυξάνει τις ανάγκες που υπάρχουν. Είναι σε στασιμότητα η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και δεν θα πρέπει να μειωθούν έτσι περαιτέρω οι πιστώσεις. Ο λόγος για τον οποίο εμείς κάνουμε τις προτάσεις αυτές είναι σαφής. Η πολιτική συνοχής δεν θα πρέπει να είναι μία απλή, ένας απλός κατεωνισμός πιστώσεων δεξιά και αριστερά, αλλά μία ριζοσπαστική πολιτική ανανέωσης των περιφερειών. Κάτι το οποίο θα μπορέσει να αλλάξει το ίδιο του το νόημα και μερικές φορές οι παρεμβάσεις της Ένωσης γνωρίζετε ότι αντιμετωπίζονται με αρνητικό τρόπο. Περισσότερο από το παρελθόν λοιπόν θα πρέπει να συνδέσουμε την πολιτική μας αυτή με το σύνολο της προβληματικής διακυβέρνησης οικονομικής της Ένωσης. Σαν παράδειγμα, η συζήτηση που θέτει σε αντίθεση τα χρηματοδοτικά υπάρχοντα μέσα με αυτά που προβλέπονται από το σχέδιο Juncker δεν είναι καθόλου χρήσιμη. Κινδυνεύουν να καταργήσουν την πολιτική σύνοχης ή να την μειώσουν ακόμα περισσότερο, υποκαθιστώντας τα αποχρηματοδοτικά μέσα, τα οποία έχουν το ελάττωμα να συγκεντρώνονται κυρίως στις πιο πλούσιες περιοχές και συνεπώς στις λιγότερο περιφερικές. Τα μέσα τα οικονομικά τα οποία στηρίζει το σχέδιο Juncker ε, βασίζονται στις ανάγκες των αγορών, αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνουν συνεισφορές και των διαφορετικών ταμείων, που είναι όμως κατά τα άλλα απαραίτητα για να πετύχουμε τους στόχους οι οποίοι συνδέονται με τα περιφερικά εδάφη και που έχουν σαν στόχο την δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την ανάπτυξη. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε κατά του σχεδίου Juncker, αλλά θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα μέσα που έχει στη διάθεσή του. Θέλουμε μια καινοτόμο λοιπόν αντιμετώπιση η οποία να κάνει τις περιφέρειες να συμμετέχουν περισσότερο και να συντονίσουμε τις παρεμβάσεις αυτές από κοινού σε μια πολυετή βάση προγραμματισμού για να διασφαλίσουμε στις περιφέρειές μας ε, μια ουσιαστική ανάπτυξη. Πάνω σε αυτό το θέμα νομίζω ότι οι περιφέρειές μας θα πρέπει να κάνουν προτάσεις και ζητάμε ένα πεδίο, ε, μια πλατφόρμα συζήτησης και συντονισμού έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη διάδραση ανάμεσα στις συνεισφορές από τη μία και τα πολιτικά αμέσα από την άλλη. Θα μου επιτρέψετε να κάνω και μία πρόταση την οποία θεωρώ ότι μπορεί να είναι σημαντική για το μέλλον. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ερεσιμότητα εξ άντε, εκ των προτέρων. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τους πόρους με πιο επιλεκτικό τρόπο και να τους εντάξουμε σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο το οποίο να έχει μια ευρωπαϊκή πραγματικά διάσταση και όχι μόνο περιφερειακή ή εθνική μια κοινή στρατηγική αντίληψη για όλη την Ευρώπη λοιπόν, ε, αποφεύγοντας ε, να πολυδιασπάσουμε τους πόρους. Σαν παραδείγμα στη δική μου περιφέρεια θελήσαμε το περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης, το σύνολο των διαθεσίμων πόρων δηλαδή, τα οποία διαχειριζόμαστε. Θέλουμε λοιπόν το πρόγραμμα αυτό να έχει πέντε βασικούς στόχους, οι οποίοι περιλαμβάνονται και στη στρατηγική Ευρώπα 2020. Απασχόληση, έρευνα, ανάπτυξη, καταπολέμηση της φτώχειας και καταπολέμηση γενικά και των συνεπειών των κλιματολογικών αλλαγών. Νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε όλα αυτά τα μέσα να τα λάβουμε υπόψη μας, συνδυάζοντας βέβαια και τα διαθέσιμα σε περιφερειακό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να καταστήσουμε ακόμα πιο ισχυρό τον δεσμό ανάμεσα στα διαφορετικά ταμεία από τη μία και σε όλα τα υπόλοιπα από την άλλη. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή στρατηγική η οποία να προσαρμόζεται στις διαφορετικές πραγματικότητες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, δίδοντας όμως το σύνολο της Ευρώπης κάποια θετικά κίνητρα. Όπως είπα όμως μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε επίπεδο περιφερειακό. Έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε θα έλεγα την πολυδιάσπαση των ευρωπαϊκών πιστώσεων και θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε ε, την ανάπτυξη των περιφερειών μας. Δεν θα φοβόμουν να πω ότι ε, η αιρεσιμότητα η μακροοικονομική είναι κάτι το οποίο δημιουργεί προβλήματα έτσι όπως δημιουργήθηκε μέχρι τώρα. Αυτό ισχύει κυρίως για περιοχές όπως η Ισπανία και την Πορτογαλία για το 2017. Γι' αυτό λοιπόν οι αλλαγές οι οποίες έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θετικές. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όμως. Οι περιφέρειες δεν έχουν ευθύνε για τους κανόνες τους οποίους επιβάλλει το Σύμφωνο Σταθερότητας. Και γι' αυτό θα ήταν παράλογο και οικονομικά και πολιτικά να τιμωρηθούν οι περιφέρειες γιατί δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προκαλέσει την παραβίαση των κανόνων. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά στους τοπικούς πληθυσμούς. Οπότε λοιπόν θα έφεται σε δυσκολία την Ευρωπαϊκή Ένωση την οποία για μια ακόμη φορά θα βλέπαμε σαν μια γραφειοκρατική πραγματικότητα η οποία επιβάλλει την λιτότητα και τους αυστηρούς κανόνες μόνον. Στη δική μου περιφέρεια και μπορώ να σας διαβεβαιώσω και αυτό ισχύει και για άλλες περιφέρειες ότι έχουμε πετύχει πολλά σε επίπεδο εξυγχρονισμού, σε επίπεδο εξοραϊσμού, σε επίπεδο δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, σε επίπεδο βοήθεια στις παραγωγικές μονάδες Όλα τα έχουμε πετύχει και χάρη στη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπαιξαν λοιπόν σημαντικότατο ρόλο για τους πολίτες τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως θα πρέπει να βρούμε μέσα έτσι ώστε αυτή η πραγματικότητα να γίνει πιο γνωστή στους πολίτες. Να το κατανοήσουν οι πολίτες. Κλείνοντας, απαιτείται να απογραφειοκρατικοποιήσουμε, ε, να απλοποιήσουμε θα πρέπει δηλαδή να μπορούμε επίσης να επαληθεύουμε με σωστό τρόπο τα αποτελέσματα των πολιτικών τις οποίες ακολουθούμε. Γι' αυτό λοιπόν το αφήγημα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να εξακολουθεί να σέβεται τους στόχους που έχουμε μέχρι τώρα και να ενισχυθεί η πολιτική συνοχή σαν βασική πολιτική για την ανάπτυξη της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρούξ έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ, να ακούσουμε την παρέμβασή σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ να σας πω πώς λέγομαι. Λέγομαι Νίκολας Μπρούξ. Είμαι διευθυντής ε, της Περιφερειακής Πολιτικής ε, στην διάσκεψη των παράκτιων περιφερειακών περιοχών και έχω έρθει εδώ για να σας παρουσιάσω σήμερα την έκβαση κάποιων εκθέσεων, μελετών μάλλον, που κάναμε στο πλαίσιο της διάσκεψης. Η πρώτη έρευνα, και πάνω σε αυτή θα επεκταθώ πιο πολύ, είναι η εδαφική διάσταση των χρηματοοικονομικών μέσων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και συνεχεία θα σας μιλήσω για δύο-τρία λεπτά για τα πορίσματα μιας άλλης μελέτης την οποία δημιουργήσαμε πέρυσι για το ρόλο των περιοχών και των εταιρικών σχέσεων, πάντα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και έχω και έντυπα, αντίτυπα στην αίθουσα, στο βάθος της αίθουσας, για όποιον ενδιαφέρεται. Στην διάσκεψη τα τελευταία δύο-τρία χρόνια προσπαθήσαμε να οικοδομήσουμε, αν θέλετε, ένα σώμα αποδείξεων για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η πολιτική συνοχή. Και μια από τι βασικέ πτυχέ που θέλαμε να μελετήσουμε είναι η χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων. Και εξετάσαμε τι υπάρχει ως βιβλιογραφία, τι ε, μελέτες και τη επιτροπής ε, Ρέγγι, αλλά είδαμε ότι δεν είχαν εξεταστεί τα ζητήματα που εμείς θέλαμε να μελετήσουμε. Πρώτο, από, αυτό, από αυτά ήταν κατά πόσον υπάρχει εδαφική διάσταση στα χρηματοοικονομικά μέσα. Αυτό είναι το πρώτο ζήτημα. Και το δεύτερο ήταν το κατά πόσον ε, τα χρηματοοικονομικά μέσα και εργαλεία είναι τα πλέον κατάλληλα μέσα για την επιτυχία των στόχων τη πολιτική συνοχή. Νωρίτερα φέτο λοιπόν ενεργήσαμε μία έρευνα ε, στα μέλη. 36 είναι οι περιοχέ, ε, οι περιφέρειες που συμμετείχαν στη μελέτη από 15 διαφορετικέ χώρε και μπορείτε να δείτε και το χάρτη. Να δείτε δηλαδή ποιες ήταν οι περιφέρειες που συμμετείχαν. Προσπαθήσαμε να καλύψουμε ε, από γεωγραφικής πλευράς και τις πιο αναπτυγμένες και τις λιγότερο και τις μεταβατικές ε, και διαφορετικά είδη περιφερειών, τις εξόγως από, κέντρες κτλ. Νομίζω ότι αυτό το οποίο προκύπτει από αυτή τη ε, μελέτη είναι κατ' ουσίαν τέσσερα μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα είναι ότι σε σχέση με τις ισχυρισμούς της ε, Κομισιόν για την αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών εργαλείων. Θα ξέρετε καλύτερα από μένα ότι στην απαρχή ε, της, της περίοδου προγραμματισμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πλασάρει αυτά τα εργαλεία ως έναν τρόπο με τον οποίο θα δημιουργηθεί απασχόληση και ανάπτυξη. Είχαν μιλήσει για μόχλευση, για ενίσχυση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στη πολιτική συνοχή και το καθεξής. Αυτό θέλησαμε να το ελέγξουμε, να το δοκιμάσουμε. Και το πρώτο μήνυμα λοιπόν που προκύπτει από την ε, μελέτη είναι ότι ναι πράγματι ήταν ε, επαληθεύθηκαν οι ισχυρισμοί της Κομισιόν, πράγματι δημιούργησαν θέσεις εργασίας, δημιούργησαν ανάπτυξη τα μέσα αυτά. Ε, βλέπετε διάφορα παραδείγματα σε αυτό το χάρτη, ΜΜΕ που ε, επιχορηγήθηκαν και στηρίχτηκαν με δάνεια, επιχορηγήσεις και τα λοιπά. Πράγματι λοιπόν δημιουργήθηκε και μόχλευση, δεν θα σας διαβάσω τα παραδείγματα, υπάρχουν κάποια εξαιρετικά παραδείγματα. Το πρώτο, που πού να το διαβάσετε βέβαια, γιατί είναι πολύ μικρά τα άραματα, τέλο πάντων είναι πολύ καλή αυτή η περίπτωση του Λαγκεντόκ Ρουσιγιό που είχαμε 5,8 ε, παραπάνω κονδύλια, μόχλευση δηλαδή από το αρχικό ποσό. Επίσης, ε, πράγματι, προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων έγινε πραγματικότητα και ιδίως εν καιρό κρίσης. Αυτό ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Όμως, το δεύτερο μήνυμα, πολύ ισχυρό και αυτό, είναι και αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο ζητήσαμε και τη γνώμη των περιφερειών σε αυτή τη μελέτη, είναι ότι τα χρηματοοικονομικά εργαλεία δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν πλήρω τι επιχορηγήσει. Για ποιο λόγο, διότι πρώτον, δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα αυτά τα εργαλεία για να στηρίξουν τα project σε όλου του εμβληματικού στόχου ε, πολιτική συνοχή. Και αν δείτε κάτω δεξιά το διάγραμμα βλέπετε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία των 23 περιφερειών που έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα εργαλεία. Βλέπετε ότι ήταν αποτελεσματικά, χρησιμοποιήθηκαν για τους θεματικούς στόχους 1, 3 και 4, δηλαδή σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, έρευνα ανάπτυξη και ενοτομία, χαμηλό άνθρακα, αλλά όχι τόσο στους άλλους θεματικούς στόχους. Αυτά είναι τα πρώτα σημεία. Ένα άλλο είναι πως μας είπαν οι περιφέρειες ότι αν ε, θέλει κανείς να χρηματοδοτήσει καινοτόμα ή υψοκίνδυνα ε, προγράμματα, μπορεί να το κάνει πιο αποτελεσματικά με τις επιδοτήσεις, με τις επιχορηγήσεις. Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία είναι καλύτερα για τη στήριξη ε, σχεδίων και έργων που είναι πολύ πιο κοντά στις αγορές, το εξήγησε και ο πρόεδρος Ρώση μόλις προηγουμένως. Κάτι άλλο που μας δίδαξε αυτή η έρευνα είναι πως τα χρηματοοικονομικά εργαλεία συνήθως δεν χρησιμοποιούνται τόσο και είναι και λιγότερα αποτελεσματικά σε περιφέρειες όπως οι λιγότερα εμπιγμένες σιωτικές περιοχές, ε, αεροκατοικημένες περιοχές, ε, ενώ λειτουργούν καλύτερα σε όριμες ανταγωνιστικές αγορές. Είδαμε επίσης Λίγε να είναι οι περιφέρειες με μικρότερα περιφερειακά προγράμματα όπως στην Ολλανδία. Εκεί αποφασίστηκε να μην χρησιμοποιηθούν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία γιατί ήταν πολύ πολύπλοκα. Και ένα άλλο ε, σημείο ήταν ο νοούμενο ε, ανταγωνισμός μεταξύ των ε, σχεδίων, εγγυήσεων και άλλων εργαλείων που υπάρχουν σε περιφερειακό επίπεδο και με αφενός αυτών και αφετέρου των μέσω της πολιτικής συνοχής των εργαλείων αυτών των χρηματοοικονομικών. Τρίτο μήνυμα. Τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία λειτουργούν ε, είναι επιτυχημένα μόνο ανάλογα με τον τύπο της περιφέρειας και στις χώρες όπου τα χρησιμοποιούν ήδη. Τέταρτο και τελευταίο μήνυμα πόσο ε, είναι πολύ απλά αυτά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Αυτό ήταν το τέταρτο μήνυμα. Ε, στην ενδιάμεση αναφέρω θα γίνουν προσπάθειες ε, να απλουστευτεί κάπως το σύστημα. Αυτή, αυτό ήταν το feedback. Υπάρχει κάποιες φορές αντίφαση στις νομοθεσίες σε εθνικό περιφερειακό επίπεδο. Τι κατευθυντές γραμμές ισχύουν για τις κρατικές νησίες, για παράδειγμα. στη χώρα των Βάσκων, Πέντε Λαλουάρ, χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιήθηκαν μάλλον αυτά τα εργαλεία στις προηγούμενες περιόδους, αλλά για τους λόγους που ανέφερα δεν αποφάσισαν να τα χρησιμοποιήσουν αυτή τη φορά. Άλλε περιφέρειε είπαν ότι τα κριτήρια πλεξιμότητας είναι πολύ στενά για τα προσχρηματοδότηση σχέδια και αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα. τέλο σαφές από την έρευνα ήταν το ότι το επίπεδο διοικητικής ικανότητας, ε, εμπειρίας ποικίλει σημαντικά από τη μια περιφέρεια στην άλλη. Είδαμε επίση ότι οι περιφέρειες οποίες χρησιμοποιούν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία στην τελευταία περίοδο τα ξαναχρησιμοποιούν γιατί έχουν αποκτήσει εμπειρία με την όλη αυτή διαδικασία. Για να ολοκληρώσω λοιπόν. Το πρώτο τμήμα της παρουσίασής μου είναι κάποιες συστάσεις που θέλω να σας ε, διατυπώσω, οι οποίες προέκυψαν από αυτό ή την ε, Το είπε και ο πρόεδρος ε, Παροδό, ο πρόεδρος Ρώση. Με βάση τα πρόσφατα αυτής της έρευνας, η πολιτική συνοχή στο μέλλον πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνδυάζει τις επιχορηγήσεις με τα χρηματοδομικά εργαλεία. Υπάρχουν στόχοι, αποστολέ που σίγουρα ε, είναι πολύ καλύτερα προσαρμοσμένε για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία, άλλε για τι ε, επιχορηγήσει. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η αύξηση τη χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων δεν γίνεται με το σωστό τρόπο. Δεν θα πρέπει να είναι αυτό ο σκοπός. Τα είπε και ο πρόεδρο Ρώση. Και περισσότερη ευελιξία είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. Ευελιξία για την νομοθεσία. Να σας δώσω τώρα κάποια άλλα στοιχεία σε ό,τι αφορά τη δεύτερη μελέτη για το ρόλο των περιφερειών και εταιρικών σχέσεων, φωνών εταιρικής σχέσης ε, για την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Εκεί είδαμε το διαβόητο άρθρο 5 και θέλαμε να ελέγξουμε και το πραγματικό επίπεδο συμμετοχής των περιφερειών στην πολιτική συνοχής. Πήραμε περίπου 40 απαντήσει ε, από περιφέρειες από 16 διαφορετικά κράτη-μέλη. Βλέπετε λοιπόν εδώ τον, κατά, την, τον Άτλαντα. Πολλές και διάφορες ε, περιφέρειες. Ε, βλέπετε και το επίπεδο ευθύνης, το επίπεδο ευθύνης των περιφερειών στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Θεωρούσαμε ότι δεν υπήρξε συσχέτιση μεταξύ του επίπεδου αποκέντρωσης, περιφερειοποίησης αφενός και του επίπεδου ευθυνών αρμοδιοτήτων που έχουν οι περιφέρειες στις χώρες αυτές. Για την Ισπανία, για παράδειγμα, βλέπετε ότι κάποιες περιφέρειες είναι ένα είδος ενδιάμεσου φορέα διαστατικού ταμείου, παρότι υπάρχουν πολλές περιφερειακέ αρμοδιότητες στην Ισπανία και από την άλλη πλευρά βλέπουμε σε κάποια νησιά διαφορετικά αποτελέσματα. Να σας δώσω και εδώ κάποια βασικά πορίσματα. Για το άρθρο θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία από τις ε, περιφέρειες. Περισσότερες είπαν ότι συμμετέχουν. Εμείς τι είδαμε όμως. Είδαμε ότι υπάρχει μια διαφορά. Άλλο συμμετέχω, άλλο είμαι υπεύθυνο για τη διαχείριση των κονδυλίων. Και από τη μελέτη ε, προέκυψε πως αυτό εν μέρει οφείλεται στην αοριστία, στην ασάφεια της διατύπωσης ε, του ΣΥΠΕΡ και του άρθρου 5 Δηλαδή, ναι, ωραία, εκπληρώσαν όλε τι απαιτήσει του άρθρου 5 κτλ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι συμμετέχουν περιφέρειες ε, και πολύ ενεργά. Ένα άλλο είναι ότι και για την περίοδο των νησιών. Το άρθρο 174 δεν είχε ως αποτέλεσμα να ληφθούν ιδιαίτερως υπόψη αυτές οι περιφέρειες. Εδώ βλέπετε τη συσχέτιση μεταξύ των θεματικών στόχων ε, της πολιτικής συνοχής και των επιπέδων ε, αρμοδιοτήτων ευθυνών. Το συμπέρασμα εδώ είναι λοιπόν ότι ακόμα και σε ουδέτερα κάπως ε, κράτη, σε διοικητικό επίπεδο υπάρχει μια, μια συνεργασία σε όλα τα σε θεματικούς στόχους. Ολοκληρώνοντας κάποιες συστάσεις πιο ποιοτικέ θα ήταν εταιρικέ σχέσεις, αν το άρθρο 5 ήταν πιο ισχυρό ε, και εφαρμοζόταν καλύτερα. Και ένας από τους τρόπους για να το εγγυηθούμε αυτό, την ποιοτική εταιρική σχέση δηλαδή, είναι περισσότερες ευθύνες και αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα είναι έτσι ένας αποτελεσματικός θεματοφύλακας ε, των αρχών της πολιτικής συνοχής. Τέλος. Οι νησιωτικές περιοχές θα πρέπει να τύχουν ειδική ε, μεταχείρισης ε, και τους δοθεί ξεχωριστή σημασία, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπρούξ. Ζητούμε συγγνώμη. Ξέρω, είμαι πολύ κακή στα ονόματα. Σας είχα αποκαλέσει μπρόκες πριν. Συνεχίζουμε τώρα με τη συζήτησή μας. Η κυρία Μπρέντσα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Ρώση για τις πληροφορίες που μας έδωσε γύρω από την πολιτική συνοχής και οι οποίες πράγματι τείνουν, θα έλεγα στον ίδιο ορίζοντα με το δικό μας. Η Επιτροπή μας έχει ήδη αρχίσει να επεξεργάζεται τις προτάσεις αυτές και νομίζω ότι αυτά που μας είπε ο Ρώση θα βοηθήσουν για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Να κάνω κάποιες σκέψεις, να εκφράσω κάποιες σκέψεις για ορισμένα από τα στοιχεία που μας έδωσε ο Ρώση. Η πολιτική συνοχής έχει νόημα εφόσον αφορά όλες τις περιφέρειες. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του 2014 μας λέγουν ότι η διαφορά ανάμεσα στις περιφερικές περιοχές με τις κεντρικές παραμένει αλλά ε, πολλές περιοχές στο κέντρο της Ευρώπης ε, κατά τη διάρκεια της τελευταίας περίοδου, με ελάχιστες δυστυχώς εξαιρέσεις, έχουν ε, υποστεί τα αρνητικά αποτελέσματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Συνεπώς, οι επενδυτικές δυνατότητες μειώθηκαν και η πολιτική θα πρέπει να είναι μια πολιτική που θα βοηθήσει όλες τις περιφέρειες να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό με τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί πράγματι η Ευρώπη ως προς αυτό έχει πολλά να κάνει. Δεύτερον, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Ρώση, η ανάγκη απλούστευσης, απλοποίησης. Είναι κάτι το οποίο αισθάνονται όλοι θα έλεγα στον τομέα αυτό. Και οι προτάσεις οι οποίες γίνονται θα πρέπει να εφαρμοστούν σε κάποια φάση έτσι ώστε να περάσουμε στην απογραφή ε, ε, ε, να να μην είναι πλέον τόσο γραφειοκρατικές οι καταστάσεις και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε σωστά τις ανάγκες τις οποίες έχουν και οι διαχειριστές των πιστώσεων αυτών σε επίπεδο πρακτικό. Θα ήθελα να μου πει ο πρόεδρος Ρώση πώς αντιμετωπίζει ένα θέμα το οποίο μας έχει ήδη απασχολήσει, το θέμα των συνεργειών, όχι ε, συγχύσεων και όχι αντικαταστάσεων, αλλά συνέργεια ανάμεσα στο ΕΦΣΙ, το στρατηγικό δηλαδή ταμείο, και τις πολιτικές ε, συνοχής. Εμείς λοιπόν έχουμε από τη μία κάνει προσπάθειες έτσι ώστε τα ταμείο Ιούνκερ να μπορέσει να επηρεάσει το σύνολο του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Υπήρου, του, Ευρωπαϊκ, του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καλό θα είναι να αρθούμε σε αυτά τα οποία μας έλεγε ο κύριος Μπρούξ προηγουμένως, το σχέδιο Juncker να μπορέσει να υποστηρίξει και σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες όμως να γίνονται αντικείμενο συντονισμού σε επίπεδο περιφερειών με παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασωθούν κάποια τμήματα της αγοράς τα οποία δεν μπορούν να βρουν τους απαραίτητους αν θέλετε τρόπους να το κάνουν μέσω ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων. Πώς βλέπετε λοιπόν με συγκεκριμένο τρόπο την συνέργεια που θα πρέπει να υπάρξει ανάμεσα στα ταμεία συνοχής, στα χρήματα, στις πιστώσεις του Ταμείου Συνοχής ε, και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε για μεγάλα προγράμματα, ε, να χρησιμοποιήσουμε ε, τα χρήματα του Στρατηγικού Ταμείου. Για τα επιτόπου, αν θέλετε, μικρότερα προγράμματα το Ταμείο Συνοχής και για τα μεγαλύτερα και ευρύτερα το ΕΦΣΥ. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό. Πιστεύετε ότι συγκεκριμένα η συνέργεια αυτή μπορεί να επιτευχθεί, γιατί μέχρι τώρα δεν το έχουμε κάνει. Είναι ελάχιστες οι δυνατότητες πραγματικής συνέργειας, αν θέλετε. Να δούμε λοιπόν αν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. και πάνω σε αυτό τι συμβουλές μπορείτε να μας δώσετε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάκοφτσης έχει το λόγο. Επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω έναν παλιό φίλο, τον κύριο Ρώση, τον είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με εξαιρετικό τρόπο μαζί του όταν ήμουν αντινομάρχης της Ίστρια. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω εδώ. Εξ αρχής θα ήθελα να πω κάτι. Το ανέφερα πολλές φορές εδώ. Άφησα την καρδιά μου στην Ίστρια, στο περιφερειακό επίπεδο, παρότι έχω την τιμή να είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό και από την αρχή θα ήθελα να μοιραστώ όλες τις ανησυχίες που εξέφρασε ο κύριος Ρώση στην παρουσίασή του. Ανέφερε το γεγονός πως ο κύριος Γιούγκερ δεν ανέφερε την πολιτική συνοχής και την περιφερειακή πολιτική στην κατάσταση της Ένωσης. Εγώ πιστεύω πως αυτό δεν έγινε κατά λάθο. Δεν είμαι σίγουρη εάν μετά, σίγουρο αν μετά το 2020 θα έχουμε μια καλύτερη περιφερειακή πολιτική και πολιτική συνοχής ή καλύτερα περιφερειακά και διαρθρωτικά ταμεία. Κατά την άποψή μου κινούμαστε προς μια διαφορετική κατεύθυνση και η πτυχή της ανάπτυξης του περιφερειακού επίπεδου έχει δεύτερη προτεραιότητα. Οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για αυτό το λόγο θα ήθελα να υποστηρίξω τον κύριο Ρώση και τη διάσκεψη παράκτιων περιφερειακών περιοχών της Ευρώπης, της οποίας μέλος ήμουν. Θα ήθελα να συζητήσω με την κυβέρνησή σας για να ενδυναμώσουμε την πολιτική συνοχή αν θέλουμε να διατηρήσουμε τον ρόλο της στο επίπεδο που έχει σήμερα. Είμαι πεπισμένος πως η αρχή της επικουρικότητας που είναι παρούσα στη συνθήκη της Λισαβόνας αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την υλοποίησή της, κατά την της, θα γίνει σεβαστή. Επίσης θα ήθελα να πω το εξής. Συμφωνώ πως το σύμφωνο σταθερότητας δεν θα πρέπει να περιέχει κυρώσεις. Δεν ήθελα να αναφέρω χτε κάποιε λεπτομέρειε, αλλά είχαμε μια συζήτηση με υπουργού από την Ισπανία και την Πορτογαλία με διαφορετικό σκοπό. Τώρα όμω θα ήθελα να μιλήσω, να πω κάτι. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπει κανεί συναδέλφου από την Καταλωνία και τη χώρα των Βάσκων, από την πολιτική ομάδα τη Άλντε να μην λαμβάνουν υπόψη την διακυβέρνηση της ισπανικής κυβέρνησης. Αλλά όταν ο κύριος Ρώση αναφέρεται στο θέμα, τότε έχει διαφορετική σημασία. Γι' αυτό και θα ήθελα να τονίσω πως εάν αποτύχουμε να χρηματοδοτήσουμε το περιφερειακό επίπεδο, τότε οι πολίτες θα υποφέρουν και δεν θα πρέπει να το τιμωρήσουμε γι' αυτό. Ίσως μιλάω συνέχεια για την περιφερειακή πολιτική. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Μεταξύ λόγια χαίρομαι πολύ που βλέπω τον κύριο Ρώση εδώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Μπρούξ και τον κύριο Ρώση για την παρουσία τους εδώ. Νομίζω ότι ήταν σωστά που στρέφουν την προσοχή μας στις περιφερειακές και θαλάσσιες περιοχές. Εδώ και 1,5 χρόνο ασχοληθήκαμε με τον ισιωτικό χαρακτήρα στα πλαίσια της έκθεσής μας και το κείμενο ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο τον μήνα Φεβρουάριο. Είναι ένα κείμενο το οποίο Ακριβώς σε αυτό ε, θα έλεγα υπογραμμίζει το σημείο που θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Και στα πλαίσια της συζήτησης και της ψηφοφορίας υπήρξε θα έλεγα μεγάλη στήριξη και η συζήτηση συνεχίζεται ακόμα και σήμερα και εδώ και αλλού. Είναι λοιπόν ένα σημείο συζήτησης, είναι ένα σημείο θα έλεγα προβληματισμού, καθορισμού των περιφερειών των νησιωτικών περιοχών και στον τομέα των μεταφορών, του τουρισμού, της γεωργίας. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος για να ξεπεράσουμε τα όρια τα διαρθρωτικά και τα περιβαλλοντικά, τα οποία λειτουργούν σαν τροχοπέδι στην ανάπτυξη των περιοχών αυτών και δεν μπορούμε να δώσουμε τις απαιτούμενες εγγυήσεις για την εδαφική συνοχή. Η Επιτροπή μας ΡΕΤΖΙ φυσικά το συζητά το θέμα αυτό, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα όργανα τα οποία εμπλέκονται και τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις πολιτικές αυτές, τις πολιτικές υπέρ των ε, περιφερειών. Δύο παραδείγματα σας δώσω, χωρίς να μακρηγορήσω. Έχουμε προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού για τις κρατικές βοήθειες, τις κρατικές επιδοτήσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Σικελία έχουν ξεκινήσει κάποιες διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται για τη χρηματοδότηση ας πούμε των αερολιμένων που είναι μέχρι ένα εκατομμύριο και τα οποία θα πρέπει να είναι είτε 100 χιλιόμετρα είτε μία ώρα τουλάχιστον οδήγησης διαφορά όπου από το σημείο που λειτουργεί ένας διαφορετικός αερολιμένας. Μερικές φορές αυτά τα θέματα είναι δύσκολα και πολλές φορές θα έλεγα έχουμε να κάνουμε με δυσκολίες οι οποίες ε, δύσκολα μπορεί να ξεπεραστούν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε το πώς επιτρέπεται να λειτουργούν οι κρατικές επιδοτήσεις στην περίπτωση των περιοχών των απομεμακρυσμένων και των περιφερειακών. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με την έκφραση από κοινού συμφερόντων και γι' αυτό έχουμε κάθε συμφέρον να συμπέσουν η προσπάθειά μας με τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ευκαιρίες είναι πολλές. Εγώ αναφέρομαι στις μεταφορές συχνά γιατί οι μεταφορές ε, θα έλεγα φύγουν άμεσα ε, τον Ευρωπαίο πολίτη. Η κινητικότητα και η διευκόλυνση της κινητικότητας σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας. Νομίζω ότι όλα αυτά θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Νομίζω ότι και σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών από πλευράς του Δημοσίου, θα πρέπει να γίνεται μια σωστή επιλογή για τις γραμμές οι οποίες χρηματοδοτούνται και οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Η ερμηνεία των κριτηρίων αυτών και ο καθορισμός των γραμμών που επιδοτούνται δεν είναι ξεκάθαρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει στην παρούσα φάση κάποιες κατευθυντήριες γραμμές ε, και έχει ξεκινήσει και μια δημόσια διαβούλευση έτσι ώστε να ξεπεραστούν οι διαφορετικές τρευλώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να ερμηνεύσουμε τα άρθρα 15, 16 και 17 με εκτατικό τρόπο και σε σχέση με τις απομεμακρυσμένες περιοχές και σε σχέση με τις νησιωτικές περιοχές. Τώρα για να κλείσω λίγο, θα έλεγα ότι η σημασία έχει να προσπαθήσουμε να ορίσουμε σωστά το πεδίο στο οποίο θα εργαστούμε. Μας ενδιαφέρουν πεδία όπως και η γεωργία σαν παράδειγμα. Είναι σαφές ότι οι απομεμακρυσμένες περιοχές έχουν κόστος παραγωγής γεωργικών προϊόντων υψηλότερο από άλλες και γι' αυτό πρέπει να διευκολυνθούν στην εμπορία τους και τη διάθεσή τους. Όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν εξάντε πριν από το κλείσιμο του κανονισμού. Ξέρουμε ότι οι δυνατότητες που έχει η DG Regio είναι περιορισμένες. Απαιτείται λοιπόν μια ευρύτερη στρατηγική και μια ευρύτερη συζήτηση. Thank you. Thank you very much, Mr. The floor is yours. Oui, merci, madame. Euh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τους κυρίους Ρώση και Μπρούξ για τις παρεμβάσεις τους και για την ανταλλαγή αυτή απόψεων που είναι πολύ επίκαιρη, διότι τελικά οι παρεμβάσεις τους έθιξαν ζητήματα επικαιρότητα που απασχολούν και την Επιτροπή μας εδώ. Θέλω να σημειώσω καταρχάς ότι τα λόγια που ε, ακούσαμε και ιδίω ε, τα σχόλια για τις μελέτες των χρηματοοικονομικών εργαλείων ε, θα μας εμπλουτίσουν τη συζήτηση και θα βοηθήσουν τον εισηγητή Νουράκοφ στην εκπόνηση της έκθεσής του. Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση που μπορεί να γίνει, με βάση την οποία η αυξημένη προσφυγή στα χρηματοοικονομικά εργαλεία δεν θα πρέπει να είναι αυτός σκοπός, δεν θα πρέπει να είναι συστηματική, γιατί τελικά πρόκειται για κάτι που θα πρέπει να αποφασίζεται επιτόπου από τους ε, κυρίους των έργων ε, και θα εξαρτάται από τα ίδια τα έργα επιλογή του χρηματοοικονομικού εργαλείου. Εγώ νομίζω ότι και οι γαλλικές περιφέρειες ε, συμφωνούν και θα ήταν αντίθετες με έναν αυτόματο και ποσοτικοποιημένο στόχο για τη χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων. Ε, απαιτείται απλά ευελιξία και ευφία και συμπληρωματικότητα επιτόπου. Να χρησιμοποιούνται δηλαδή τα χρήσιμα ε, αφενός χρηματοοικονομικά εργαλεία και τα άλλα εργαλεία της πολιτικής συνοχής αφετέρου. Έχουμε σε ένα άλλο ζήτημα. Μια πολιτική τοποθέτηση που ακούστηκε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Έχω μια ερώτηση. Η διάσκεψη μας είπε ότι η αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής βασίζεται στο ΑΕΠ, το περιφερειακό ΑΕΠ, αυτό είναι το κριτήριο. Με αποτέλεσμα Ενδεχομένως κάποια εδάφη που έχουν μόνιμο ελάττωμα δεν θεωρούνται αυτόματα προτεραιότητες. Ερώτηση προς τους δύο προσκεκλημένους μας. Η διάσκεψη θεωρεί ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι δείκτες πλην του ΑΕΠ ή συμπληρωματικοί δείκτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Κυρία Βάνα. Äh, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Αντιπρόεδρο Ρώση και τον Διευθυντή Μπρούξ που συμμετείχαν σήμερα στις εργασίες της Επιτροπής και εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δέσμευσή σας για την περιφερειακή πολιτική στο πλαίσιο της διάσκεψης παρακτήων περιφερειακών περιοχών της Ευρώπης όπως και τη μελέτη σας που παρουσιάσατε σήμερα και τις πληροφορίες που μας δίνετε για τα χρηματοδοτικά μέσα απέναντι στα οποία έχουμε μια πολύ κριτική στάση. Προσωπικά, όπως και οι προλαλήσαντες, συμφωνούμε τα περισσότερα από αυτά που είπατε. Χρειαζόμαστε την πολιτική συνοχή, όχι μόνο για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, αλλά επίσης για την εδαφική συνοχή, αλλά επίσης επειδή ωφελεί όλες τις περιφέρειες. Και επειδή είδαμε πως σε κάποιες περιοχ... περιφέρειες είναι η μόνη μορφή δημόσιων επενδύσεων που έχει απομείνει. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε μία υποβάθμιση αλλά μία αναβάθμιση της πολιτικής συνοχής. Ο Προλαλήσατας ζήτησε σε μια καλύτερη πολιτική συνοχή και αυτό ακριβώ είναι. Έχετε μία πρόταση με τη μείωση του γραφειοκρατικού άχθους. Πιστεύω ότι η διαφάνεια είναι επίσης ένα στοιχείο ακόμα για μια καλύτερη πολιτική συνοχής. Αλλά εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το εξής. Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις επί του παρόντος είναι η αλλαγή παραδείγματος στην επενδυτική πολιτική, την οποία θα ονομάσω πραγματικό κίνδυνο για την πολιτική συνοχής. Καθώς μειώνονται συνεχώς κονδύλια χωρίς όριο για το νέο σχέδιο Juncker που λειτουργεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Όλα αυτά δηλαδή που καταγράψατε ως κεκτημένα της πολιτικής συνοχής όπως είναι η Ευρώπη 2020, η αρχή της εταιρικής σχέσης. Όλα αυτά δεν περιέχονται εκεί. Γι' αυτό και η ερώτησή μου προς εσάς. Πώς βλέπετε τις προκλήσεις εδώ υπό το πρίσμα της αλλαγής παραδείγματος αυτού. Τι πρέπει να συμβεί ως προς το περιεχόμενο αλλά και διαρθρωτικά για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η μορφή πολιτικής αλλά και η συμπλήρωσή τους των δύο μέσων αυτών και να λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η πολιτική συνοχής να μην χάσει το χαρακτήρα αλληλεγγύης της. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζέλερ, έχει τον λόγο. Ο κύριος Ζέλερ, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ επίσης τους προλαλήσαντες και για τις εκθέσεις τις οποίες δυστυχώς έλαβα σήμερα μόλις. Δυστυχώς θα ήθελα να τις έχω μελετήσει πιο πριν. Η εντύπωση που δώσατε είναι προς σύμφωνα με τις νεότερες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο ρόλος της πολιτικής συνοχής δεν είναι πια τόσο μεγάλος. Έχετε δίκιο. Πριν από μερικά χρόνια τα διαφορετικά ταμεία ακόμα εκτιμούνταν ως το καλύτερο μέσο που μας διατίθεται. Ούτε καν γίνεται λόγος πλέον γι' αυτό. Γι' αυτό και πιστεύω πως ήρθε ο καιρός να μιλήσουμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Στην έκτη έκθεση συνοχής ο ένας πιλότας, πυλώνας της πολιτικής αυτής, όπως τη θεωρώ εγώ, δηλαδή η διασυνοριακή συνεργασία, πλέον δεν υπήρχε. Έχω μία ερώτηση. Πιστεύω πως κατάλαβα σωστά πως τα χρηματοδοτικά μέσα χαίρουν της εκτίμησής σας. Οπότε θα με ενδιαφέρε ποια κράτη εξετάσατε και σε ποιο χρονικό διάστημα. Στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού είχαμε μια έκθεση για την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών μέσων την τελευταία, στο τελευταίο δημοσιονομικό πλαίσιο. Εκεί η εικόνα ήταν διαφορετική. Εκεί είδαμε πως τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές για την καταβολή χρημάτων. Χρήματα τα οποία σταθμεύονταν πολλές φορές στις τράπεζες για να αυξηθούν τα ίδια κεφάλαια αυτών. Ενώ οι μικρές και οι μεσές επιχειρήσεις που θα έπρεπε να τα λάβουν δεν τα έπαιρναν. Το οποίο με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα τα χρηματοδοτικά μέσα αυτά να χρησιμοποιούνται σε χαμηλό βαθμό. Τώρα, αν έχετε διαφορετικές εμπειρίες, πολύ θα χειρόμουν να τις ακούσουμε. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντεμάσο, έχετε το λόγο. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κυρίους κύριους Μπρουξ και Ρώση για... και να περάσω στις ερωτήσεις. Καταρχάς, η πολυδιάσπαση των ταμείων των διαρθρωτικών Πραγματικά υπάρχουν και πάρα πολλά εμπόδια γραφειοκρατικά που δεν επιτρέπουν να υπάρξει και σωστή χρήση των χρημάτων αυτών. Υπήρξε από πλευράς του κύριου Γιούνκερ πρόταση για μεγαλύτερη ευελιξία και ελαστικότητα, αλλά κυρίως για το εύση, όχι για τα υπόλοιπα ταμεία. Και τώρα για τη μακροερεσιμότητα. Θα συμφωνήσει μαζί μας και ο κύριος Ρώση και ε, οι υπόλοιποι συνάδελφοι για να ζητήσουμε την αναθεώρηση του άρθρου 23 την κατάργηση δηλαδή της υποχρέωσης σύμφωνα με κάποιες ερμηνείες της πρότασης διακοπής των λειτουργικών προγραμμάτων για χώρες που δεν ακολούθησαν πλήρως τις συστάσεις του Συμβουλίου. Και τέλος για την ολοκληρωμένη ε, από κοινού χρήση στα πλαίσια του Horizon 2020 του ταμείου αυτού με τα υπόλοιπα ταμεία. Εσείς σκοπεύετε να ακολουθήσετε την κατεύθυνση αυτή κύριε Ρώση. Από τον κύριο Μπρουξ έχουν υπάρξει μελέτες σε σχέση με τα χρηματοδοτικά μέσα και τις περιφέρειες μπορούμε να μιλήσουμε για τις πραγματικές διαφορές ανάμεσα στις πιο ολοκληρωμένες ε, περιοχές και αυτές οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο ανάπτυξης. Υπάρχουν διαφορές στις επιδόσεις ε, των χρηματοδοτικών μέσων σε αυτές τις δύο διαφορετικού τύπου περιφέρειες. Μάλετιτς. Και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τους ε, προσκεκλημένους μας για την παρουσίασή τους, τον κύριο Μπρουξ και τον κύριο Ρώση. Θα συμφωνήσω επίσης και μαζί σας και με τους άλλους συναδέλφους ότι έχουν υπάρξει αρκετές καινοτομίες που προβλέπονται για την περίοδο 14-20, θεματολογική συγκέντρωση, καλύτερος προσανατολισμός, καλύτερος συντονισμός με την οικονομική πολιτική, ε, συσχετισμός καλύτερος των προτεραιοτήτων με τις επιτόπου περιφερειακές ανάγκες και καλύτεροι τρόποι εφαρμογής. Έχουμε επίσης πολλά μέσα τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα όπως θα έπρεπε και πολλά είναι τα κρατημέλη και οι περιφέρειες οι οποίες προσπαθούν να αποφύγουν τη χρήση τους, αν και θεωρητικά θα είχαν να κερδίσουν. Την τελευταία φορά αναφερθήκατε ε, στο λεγόμενο Simplified Cost Options, στις απλοποιημένες επιλογές κόστους. Κι όμως, ε, ακόμα και σήμερα, οι διαχειριστικές αρχές στις περιφέρειες δεν χρησιμοποιούν τις μεθόδους αυτές. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα πρέπει να εργαστούμε ακόμα περισσότερο και καλύτερα για την εφαρμογή των μέτρων που έχουν πλέον εισαχθεί. Αναφερθήκατε και στην αρχή της εταιρικότητας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο θα εμπλέξουμε περιφέρειες περισσότερο από ό,τι σήμερα να πάρουν μέρος λοιπόν στον καθορισμό των λειτουργικών προγραμμάτων. Και τι πιστεύετε τώρα για μια ιδέα που κυκλοφορεί για το μέλλον η πολιτική συνοχής να έχει ένα περιφερειακό γραφείο σε κάθε χώρα και να καταργηθούν οι δυνατότητες να υπάρχουν εθνικά, να υπάρχουν περιφερειακές μάλλον έδρες και όχι εθνικοί. Ο κύριος Μπούντα, ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο μιλητές για τις παρουσιάσεις οι οποίες κατά την άποψή μου επιβεβαιώνουν αυτό που σε ένα βαθμό ήδη γνωρίζαμε. Ότι δηλαδή η πολιτική συνοχή έχει θετικές ε, επιπτώσεις, θετικά αποτελέσματα. Βέβαια, δυστυχώς αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην καταλαβαίνει την πραγματική αξία της πολιτικής συνοχής. Προσπαθεί λοιπόν να σχεδιάσει μια πολιτική που δεν θα μπορεί πλέον να, επιτύχει τους στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε. Δεν μπορεί να πετύχουμε τους στόχους μας αν δεν έχουμε μια καλά διαρθρωμένη πολιτική συνοχής. Οι ανάγκες ε, των περιφερειών υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα. Πρέπει να μιλάμε πλέον για περιφερειακές ανάγκες και η κατάσταση δυστυχώς που έχουμε σήμερα προκαλείται από την ανικανότητα της Κομισιόν να κάνει πιο ορατή την ε, πολιτική συνοχή. Και τώρα έρχομαι στο ερώτημα θέλω να θέσω. Υπάρχουν πράγματι κάποια απορίσματα που δείχνουν ε, την προστέμενη αξία για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για οικονομική αξία κτλ. κτλ. Αν ήξερε η γνώμη ότι υπάρχει αυτή η προστέμενη αξία της περιφέρειες και αν μάθαινε ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση αυτή η προστέμενη αξία, διότι ξέρουμε και το Brexit, ποιοι ψήφισαν υπέρ του Brexit, εκεί ακριβώς που δεν... Εκεί που είχαν μάλλον δοθεί τα περισσότερα κονδύλια, εκεί ψήφισαν όμως κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα Μήπως πρέπει να δώσουμε έμφαση στην ανάγκη να είναι πιο ορατή η πολιτική συνοχή. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε στις μελέτες αυτές, τις έρευνες, είδατε, προσπαθήσατε να διαπιστώσετε πόσο ενήμερη είναι η κοινή γνώμη για την πολιτική συνοχή. Ευχαριστώ. Πρόεδρο τελευταίο. μου της κ. Φανίστελ Ροϊ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη διάσκεψη Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και επικοδομητική αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Στον κύριο Ρώση στρέφομαι. Κύριε Ρώση, είπατε να παραμείνει εκ των προτέρων αιρεσιμότητα, εξειδίκευση, θεματική κτλ. Αλλά λέτε στο μέλλον να συνδυαστεί αυτό και με μια πιο κεντρική προσέγγιση. Μιλάμε τώρα για κάτι επαναστατικό, έτσι. Κοινή διαχείριση τελικά σε επίπεδο κρατών μελών ή όπως προβλέπει η έκθεση της Προέδρου μας, εδαφική συνοχή, δυσνορική συνεργασία, εδαφική συνεργασία, να τριπλασιαστεί, να δεκαπλασιαστεί. Τα σκέφτεστε και αυτά. Δεν ξέρω, αυτό μου φάνηκε πολύ καινοφανέ ε, που είπατε. Ένα πιο γενικό ερώτημα και με βάση και τα όσα ακούστηκα στη συζήτηση, η συνοχή. Δεν φαίνεται να υπάρχει και πρόβλημα στην πολιτική αυτή. Σε δύο-τρία χρόνια θα επανέλθει η πολιτική συνοχή στο επίκεντρο ότι έχουμε κάποιες χειρότερες δυνάμεις, αλλά τελικά μόνο διαφορετικά μπορούμε να λειτουργήσουμε και γι' αυτό θα επανέλθει η συνοχή στο επίκεντρο στο μέλλον. Περιφέρειες είναι στο επίκεντρο αυτής της ανάπτυξης. Μην απελπιζόμαστε λοιπόν με το τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τώρα έχουν ένα άλλο αγαπημένο παιδί στην Κομισιόν, το ΕΦΣΙ. Εκείνη το ερώτημα τώρα. Τι θα το κάνουν αυτό το εύση. Έκλεισε τα, το ένα έτος. Πώς γίνεται όμως αυτό το πρόγραμμα να ε, ευημερίσει. Παίρνουμε σαν να έχουμε ένα γλυκό και παίρνουμε ένα φρούτο από εδώ, παίρνουμε ένα φρούτο από εκεί. Δεν υπάρχει όμως κάποια διασύνδεση με άλλα προγράμματα εκπαίδευσης ε, κτλ δεν δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να δουλέψουν αλλού, ναι. η υποδομές, στέγας κτλ. Άρα κάνουμε έτσι κατακαιρματισμένα πράγματα. Υπάρχει αυτή η πολυδιάσπαση που είπατε και εσείς. Τώρα θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τη νέα φάση, τη νέα στρατηγική μετά το 2020. Μήπως θα έπρεπε να τα πούμε πιο έξω από τα δόντια τα πράγματα. σε σχέση με το τι γίνεται τώρα. Τελευταία παρατήρηση. Γενική παρατήρηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα δεν έχει υποστήριξη. Το είπε και ο κύριος Μπούντα. Δεν έχει τα εργαλεία να κάνει μια καλή ε, εκστρατεία ενημέρωσης, πληροφόρησης. Μήπως πρέπει να πούμε στην Κομισιόν. Ξέρετε, υπάρχει ο λαϊκισμός, υπάρχει εθνικισμός, ε, τα έχετε βγει εκτός παιχνιδιού. Δεν πρέπει κάτι να κάνετε. Οι πολίτες μας, ξέρετε σε πόσο ποσοστό γνωρίζουν την πολιτική συνοχή, 30%. Πόσοι γνωρίζουν το έύση. Σε ποιον αρέσουν τα τραπεζικά κτλ. Εντάξει, οι τραπέζες έχουν τις δικές τους ε, επιδιώξεις. Οι πολίτες ξέρουν τι είναι το εύση. Άρα πρέπει να είμαστε πιο εφάνταστοι και δημιουργικοί και στις επενδύσεις. Σε ποιο θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε στα διαφορετικά πράγματα. Πολιτική συνοχή, ΕΦΣ και τα λοιπά. Πώς δεν μπορέσουμε να το πλασάρουμε με επιτυχημένο τρόπο, για πείτε μας. Να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κυρία Αντεπανάιτε. Thank you very much. Good Καλό απόγευμα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω πως έλαβα γνώση και πως θα ενημερώσω το συνάδελφο. Προσωπικά είμαι αρμόδιος για το αρμόδια για το φάκελο των εταιρικών σχέσεων και ήδη αναλύσαμε διεξοδικά τα ευρήματα της μελέτης αυτής καθώς υπάρχουν εδώ και κάποιο καιρό. Εμείς από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την υλοποίηση της αρχής της εταιρικής σχέσης συνεχίζουμε να το παρακολουθούμε διεξοδικά στο πλαίσιο των συζητήσεων με τα κράτη-μέλη. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης και όσον αφορά τη συνεργασία με εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε σύναψη τον διαφορεμένο διάλογο με τους εταίρους. Συναντιόμαστε δύο φορές το χρόνο και συζητούμε θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τις τρεις κατηγορίες εταίρων που συμμετέχουν στην ομάδα μας. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού κοινών διατάξεων. Δηλαδή τοπικές και περιφερειακές αρχές, η κοινωνία των πολιτών. Η, η επόμενη συνάντηση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, την Τρίτη. Και η συγκεκριμένη συνάντηση αυτή, η συνεδρίαση αυτή, θα εστιάσει στα βήματα προετοιμασίας για την πολιτική μετά το 2020 και οτιδήποτε που θα οδηγήσει σε μια ύστερη αργότερη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την, για την πολιτική συνοχή μετά το 2020. Ο συνήθως το Κοινοβούλιο θα υποβάλει την έκθεσή του η Επιτροπή μάλλον για να την λάβετε υπόψη. Ευχαριστώ. Κύριε Ρώση, κύριε Μπρούξ, πολλές ερωτήσεις Θέλετε να απαντήσετε ποιος θα είναι πρώτος. Ο κύριος Ρώση, εντάξει. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές που πήραν μέρος στη συζήτηση. Ήταν ιδιαίτερα σημαντικές οι παρεμβάσεις τους. Πολλά από αυτά που είπαν μπορώ να τα μοιραστώ κάλλιστα. Νομίζω ότι υπήρξε μια πλήρης επιβεβαίωση της ανάγκης να ε, επανεκκινήσουν οι πολιτικές συνοχής για μετά το 2020. Η πρώτη φάση είναι να δούμε ακριβώς πώς έχουν πάει ε, μέχρι τώρα. Νομίζω ότι για μας είναι μια δύσκολη φάση αυτή. Ο έλεγχος, η αξιολόγηση θα πρέπει να πάει καλά αν θέλουμε να ζητήσουμε την συνέχεια εφαρμογή τους. Θα πρέπει λοιπόν μετά την επταετία να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Θέλουμε επίσης να υπερασπιστούμε τις μορφές χρηματοδότησης που έχουν ήδη προβλεφθεί στα πλαίσια της συνοχής και γι' αυτό ακριβώς και η δική σας φωνή όπως είπε και η κυρία Νταμάτο και άλλοι συναδελφοί σας γιατί πράγματι από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής να μην αφαιρεθούν πόροι για να δοθούν σε άλλου είδους πολιτικές. Ε, έτσι θα αποτύχει η πολιτική συνοχής ε, εφόσον της αφαιρεθεί σιγά σιγά ο χυμός και χρησιμοποιηθεί αλλού. Τώρα κάποιες άλλες συνθετικού τύπου απαντήσεις. Πρώτον, να επιβεβαιώσω ότι έχουμε ανάγκη της πολιτικής συνοχής και δεν πρέπει να μειωθούν οι πιστώσεις τους. Δεύτερο σημείο, πολύ σημαντικό, θα πρέπει η εθνική συγχρηματοδότηση και περιφερειακή συγχρηματοδότηση να γίνεται δεκτή, να αφαιρεθεί ουσιαστικά δηλαδή από το ε, σύμφωνο σταθερότητας. Γιατί αλλιώς θα υπάρξουν πάρα πολλά προβλήματα στις περιφέρειες και δυστυχώς η πολιτική συνοχής δεν θα έχει κάποια επιτυχία. Είναι ένα αίτημα το οποίο το κάνει και το κόμμα μου και όλες οι περιφέρειες στην Ιταλία και νομίζω ότι το κάνουν το ίδιο πράγμα όλες οι περιφέρειες της RPM. Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούμε να δαπανίσουμε μερικές φορές τα χρήματα αυτά είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις γιατί μας εμποδίζει το σύμφωνο σταθερότητας. Για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το πρόβλημα. Για την το σκάνει 80 εκατομμύρια το χρόνο, 80 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ε, εμείς χρησιμοποιούμε για την συγχρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής μπορούμε να τα έχουμε στη διάθεσή μας για να επενδύσουμε, να τα επενδύσουμε, όχι να τα βάλουμε στους τρέχοντες λογαριασμούς. Να μην τα κρύψουμε δεξιά-αριστερά, αλλά να τα επενδύσουμε. Αλλά δυστυχώς τα χάνουμε διότι μας εμποδίζει να τα χρησιμοποιήσουμε ε, το ε, Σύμφωνο Σταθερότητας. Επίσης οι καθυστερήσει στη χρηματοδότηση οφείλεται στο ότι θα πρέπει να μπορούμε να αφαιρέσουμε τις συγχρηματοδοτήσεις από το Σύμφωνο Σταθερότητας. 80 εκατομμύρια για τη δική μου περιφέρεια. Καταλαβαίνετε σε στάδιο επταετίας τι σημαίνει κάτι τέτοιο, μόνο για την Τοσκάνη. Δεύτερον, θα πρέπει να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες γιατί και αυτές προκαλούν καθυστερήσεις. Οι πιο σημαντικές χρηματοδοτήσεις της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να υφίστανται τις διαδικασίες που ισχύουν και για τις κρατικές επιδοτήσεις. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει και για το σχέδιο Juncker, για το πρόγραμμα Juncker. Είναι μια διαδικασία η οποία μας δημιουργεί εμπόδια, μας δημιουργεί ανασφάλεια και η συνάδελφός σας από την Κατάνια το έθεσε το πρόβλημα και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη Σικελία αλλά για, όλες τις, για όλη τη χώρα, την Ιταλία εννοώ, αλλά και για άλλες περιφέρειες παραθαλάσσιες και περιφερειακές. Πέραν αυτού, για την μακροαιρεσιμότητα είναι προφανές ότι θα πρέπει να ζητήσουμε να μην υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες ε, δεν θα έχουν καμία επιτυχία τελικά, θα δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. Και θα ήθελα να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες περαιτέρω προτάσεις, οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την ανανέωση του τρόπου χρήσης ε, των ε, διαρθρωτικών ταμείων και να υπάρχει η δυνατότητα ενός μπόνους όταν τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Επίσης υπάρχει ο κίνδυνος της πολυδιάσπασης. Είναι αν θέλετε το πιο αδύναμο σημείο ε, του Ταμείου Συνοχής. Σε πάρα πολλές περιφέρειες και σε περιοχές γενικότερα σημειώνονται καθυστερήσεις σημαντικές λόγω της πολυδιάσπασης των πιστώσεων. Πρέπει να καταστούν πιο συνεκτικοί οι στόχοι της στρατηγικής 2020 και οι τρόποι χρήσης των διαφορετικών ταμείων. Αυτό τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε στα διαφορετικά ταμεία και στα ταμεία σύνοχης ένα πιο θεσμικό χαρακτήρα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρξουν ακόμα περισσότερα εμπόδια και καθυστερήσεις. Πρέπει όμως ε, τα διαφορετικά ταμεία να συνδεθούν καλύτερα με τη στρατηγική 2020 και θα πρέπει να αφήσουμε ελεύθερη κάθε περιφέρεια να αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα πετύχει τους βασικούς της στόχους. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα πρέπει να δώσω μια απάντηση, ίσως και κάποιες απαντήσεις, το έθεσε η κυρία Μπρέσο, αλλά και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, ξεκινώντας από τον εντοπισμό κάποιων πολύ μεγάλων προγραμμάτων, όχι ε, διασπασμένων και επιμέρους, θα πρέπει να μας υπάρξει, να μας δοθεί δυνατότητα να συνδέσουμε την χρηματοδότηση από το σχέδιο Juncker για να τα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, να συνδέσουμε τα διαφορετικά ταμεία, τη δράση τους με τη δράση του Ταμείου Juncker. Έχουμε κάνει ας πούμε πολύ μεγάλες επενδύσεις σε επίπεδο λιμενικών εγκαταστάσεων χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά ταμεία. Από μόνα τους δεν επαρκούν. Οι δημόσιες επιδετήσεις δεν επαρκούν. Κάποιες καλύπτονται από δανεισμό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια δυνατότητα σύνδεσης με το Ταμείο Juncker έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε τους στρατηγικούς στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Δεύτερον, έχουμε κάνει επενδύσεις στην κινητικότητα των αστικών περιοχών. Και εδώ πέρα από τις επενδύσεις που επιτρέπουν τα διαρθρωτικά ταμεία, καλό θα ήταν να έχουμε την δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Juncker, που είναι ε, ε, ειδικού επιτοκίου ε, δανεισμοί ουσιαστικά. Και τρίτον, υπάρχει πολιτική λογιστικής διαχείρισης που ισχύει για τις επιχειρήσεις. Καλό θα είναι να ξεκινήσουμε μια διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρησιμοποίηση του σχεδίου Juncker με τα διαρθρωτικά ταμεία τα οποία χρησιμοποιούνται ε, για τη διευκόλυνση επενδύσεων στην Ήπεθρο. Τώρα σας έδωσα τρία ειδικά παραδείγματα. Υπάρχουν πολλά άλλα. Σαν παράδειγμα σε επίπεδο καταπολέμησης της φτώχειας, σε κοινωνικά μέτρα, καταπολέμησης του αποκλεισμού, Αυτές είναι πολιτικές που μπορούν να ξεκινούν με βάση τις γενικές στρατηγικές, με βάση τις στρατηγικές της περιφέρειας, αλλά που απαιτούν εκ των υστέρων τελικά μία παρέμβαση των δυνατοτήτων του σχεδίου Juncker. που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και ε, για, ιδιωτικού, ε, για ιδιωτικές επενδύσεις αλλά και για δημόσιες. Τώρα ένας άλλος τομέας ε, βασικός είναι το Horizon 2020. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες. Μία από αυτές είναι το, η πόλη του Πιομπίνο. Έχει ενδιαφέρον. Στο Πιομπίνο συνδυάζουμε ένα λιμένα ο οποίος αντιμετώπισε μια οικονομική κρίση σοβαρή. Χρησιμοποιήσαμε ιδιωτικές επενδύσεις, διαφθορτικά ταμεία και ε, ένα σχέδιο το οποίο συνδέεται με το Horizon 2020. Λοιπόν, σε κάθε περιφέρεια μπορούμε να συνδυάσουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει βέβαια να αγνοήσουμε τις ανάγκες των πόλεων, αλλά θα μείνουμε στις περιφέρειες, θα ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική και αν για κάθε περιφέρεια εμείς σε σχέση και με τη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και σε σχέση με τις στρατηγικές 2020 μπορέσουμε να προωθήσουμε κάποια μεγάλα στρατηγικά προγράμματα για τα οποία να χρησιμοποιήσουμε όλες τις δυνατές πηγές χρηματοδότησης και το Horizon 2020 και το Ταμείο Juncker και τα Περιφερειακά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, τότε μπορούμε να έχουμε στρατηγικές επενδύσεις οι οποίες θα μας επιτρέπουν να δούμε τις ε, επιπτώσεις της χρήσης των κοινοτικών ταμείων με καλύτερο τρόπο. Κοιτάξτε δεν είναι εύκολο αυτό βέβαια, αλλά θα είναι λιγότερο γραφειοκρατικό, περισσότερο υπεύθυνο και σε σχέση με την επικοινωνία μας με τον πληθυσμό θα είναι πιο αποτελεσματικό. Τι κάνει η Ευρώπη στις περιφέρειες. Αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα, τα 7 προγράμματα, τους 5 στόχους. Είναι συγκεκριμένη η δυνατότητα της Ευρώπης να παρέμβει και θα πρέπει να φαίνεται στον κόσμο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα ήταν ένα καλύτερο, σημαντικότερο και αποτελεσματικότερο μέσο για να πετύχουμε τον γενικό στόχο τον οποίο έχουμε που είναι η ανάπτυξη. Να κλείσω, λέει ο κύριος Ρώση, ε, χαιρετώντα και τον αγαπητό φίλο Γιάκοφτσιτς για τα καλά του λόγια. Να συμφωνήσω μαζί του με την παθιασμένη υπεράσπιση από πλευράς του της πολιτικής συνοχής. Είπε ότι αν δεν περιφερειακά προγράμματα δεν χρηματοδοτηθούν θα υποφέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Όσοι έχουν περάσει από τις τοπικές αρχές ε, οι ευθύνε οι οποίες είχαν τους δείχνουν ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι σημαντικά και καθοριστικά. Και να συνεχίσω πριν τελειώσω λέγοντας ότι σε επίπεδο επικοινωνίας καλό θα ήταν, χρήσιμο θα ήταν, επαληθεύοντας αν θέλετε ε, την κατάσταση στο μέσο του χρόνου ε, της επταετίας να δούμε σε επίπεδο επικοινωνίας τι μπορεί να καταστεί υποχρεωτικό ένα τμήμα των χρηματοδοτήσεων ε, ξέρουμε ότι δεν χρησιμοποιούνται πάντα με, πιο, με τον πιο σωστό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια κατευθυντήρια γραμμή για την δημοσιοποίηση των παρεμβάσεων, της φύσης των παρεμβάσεων της πολιτικής συνοχής. Και νομίζω ότι αυτή η κατευθυντήρια γραμμή θα είναι χρήσιμη σε όλους. Thank you. Um, ευχαριστώ. Θα αρχίσω για... με το σχέδιο Juncker και την πολιτική συνοχή. Ο κύριος Ρώση ήδη έδωσε κάποια παραδείγματα για το πώς θα μπορούσαν στο μέλλον να βελτιωθούν τα πράγματα. Εγώ θέλω να επαναλάβω από την πλευρά μου ότι με, με το έγγραφό μας ασκούμε κριτική στο γεγονός ότι το ΕΦΣΙ και η πολιτική συνοχή έχουν σχεδιαστεί και αναπτύσσονται εντελώ διαφορετικά, ξεχωριστά μεταξύ του. Ε, από την Κομισιόν δεν υπάρχει ένα ισότιμο πεδίο ε, και δεν γίνεται ισότιμα η προβολή, η διαφήμιση, αν θέλετε, του ενό και του άλλου. Εμείς εστιάζουμε στους ομείς, και τα λοιπά, στις περιοχές, αλλά δεν βοηθά αυτό ε, εμάς που είμαστε φίλοι πολιτικής συνοχής. Και κάτι άλλο, και ήταν ξεκάθαρα το Κοινοβούλιο, για το οποίο σκόμε κριτική είναι η προσθετικότητα. Ποτίθεται ότι φέρνει το εύση. Δεν είμαστε σίγουροι ότι ισχύει αυτό. Γι' αυτό και στο έγγραφό μας ήμασταν ξεκάθαροι, το είπε και ο πρόεδρος Ρώση νωρίτερα. Θα πρέπει να δούμε πώς αυτά τα δύο, και το σχέδιο και την πολιτική, γιατί το ΕΦΣΙ δεν είναι παρά ένα σχέδιο. Και το σχέδιο λοιπόν αυτό, αλλά και η πολιτική, πώς μπορούν κάπως να ενοποιηθούν για τον κύριο Τσέλερ που ρώτησε για τη χρήση των χρηματοοικονομικών εργαλείων, ουσιαστικά συμφωνώ με αυτό που είπατε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, επέκρινε τη χρήση, ε, της, ε, τον τρόπο με τον οποίο είναι τη χρήση αυτών των εργαλείων. Εγώ σας έδωσα ένα παράδειγμα για το πού είχαν θετικά αποτελέσματα αυτά τα εργαλεία. Αλλά αν δείτε τη μελέτη μας, νομίζω ότι έχετε τώρα το αντίτυπο, θα δείτε ότι υπάρχει κριτική στον τρόπο τώρα που χρησιμοποιήθηκε αυτή η χρηματοδότηση. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι τα χρηματοοικονομικά εργαλεία είναι πολύ χρήσιμα, αλλά μόνο σε συγκεκριμένους θεματικούς τόπους και σε συγκεκριμένα είδη περιφερειών. Η μελέτη όμως νομίζω θα σας δώσει πιο πολλά στοιχεία, πιο πολλές απαντήσεις για την Κέντα για την επιτυχία των ε, εργαλείων αυτών σε λιγότερο αναπτυγμένες περιοχέ. Μπορείτε να διαβάσετε τη μελέτη για περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ μπορώ να σας πω ότι εξετάσαμε την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και είδαμε το εξή. Δεν έχω τώρα πάρα πολλά στοιχεία, αλλά το 71,4% της ανταγωνιστικότητας στις ε, περιοχές στόχου 2 είχαν θετική ε, άποψη και 33% μόνο στις περιφέρειες σύγκλησης. Μιλώ τώρα για τη θετική άποψη για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία και στις δύο περιπτώσεις. Άρα βλέπουμε διαφορές στις διαφορετικές κατηγορίες. Για τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα δεν θα ήταν καλύτερο, είπε κάποιο. Ναι, θα μην θα το στηρίξουμε βέβαια από πλευρά διάσκεψη ε, Αλλά να πω ότι αρχικά αυτό που θα πρέπει να γίνει είναι να πιστούν οι κύριοι Γιούγκερ και Κατάινεν για τις περιφέρειες, ότι υπάρχουν και αυτό θα ήταν το πρώτο που πρέπει να γίνει. Υπάρχουν ε, θεσμικά εμπόδια, γι' αυτό εμείς εστιάζουμε και στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βοηθήσει να γίνει σεβαστή αρχή τη εταιρική σχέση. Και έχουμε παραδείγματα στι μελέτε μα που δείχνουν ότι σε κάποια κράτη-μέλη περιφέρειε δεν εισακούστηκαν και ούτε είχαν και έναν ρόλο, μια συμμετοχή. Μπορούν να γίνουν πράγματα λοιπόν τέλος για την εκ των προτέρων αρισιμότητα ερώτηση νομίζω του κυρίου Βανίστελ Ρόι. Τα λέμε ξεκάθαρα στο έγγραφό μας. Η εξάντα αρισιμότητα από την διάσκεψή μας ε, έχει ένα συγκεκριμένο νόημα. Κάτι λέει η Κομισιόν για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που θα πρέπει να σε σχετιστεί με την πολιτική συνοχή. Εμεί πιστεύουμε ότι η σχέση υπάρχει και είναι εκ των προτέρων περιφερειακές αρχές, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκπληρώνουν πολλέ υποχρεώσει που έχουν να κάνουν με τι επενδύσει και την ανάπτυξη πριν την έναρξη των προγραμμάτων. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε για να γίνονται με συνεπή και συνεκτικό τρόπο οι επενδύσει. Σε ό,τι αφορά το... τις στρατηγικές εφιούς εξειδίκευσης, πρέπει να σα πω ότι αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό και το πιο καλό παράδειγμα εκ των προτέρων αρεσιμότητας. Μας είχαν πει όλες τις ότι ήταν εξαιρετικό το μέτρο αυτό, βοήθησε πολύ τις επενδύσεις και το βαθμολογεί θετικά και η Κομισιόν. Γιατί ενθάρρυνε τις περιφέρειες να επενδύσουν στην καινοτομία και στην έρευνα. Άρα αυτός πράγματι είναι ένας ε, τρόπος ε, να προχωρήσουμε προς τα εμπρός και εδώ θα ολοκληρώσω. Ευχαριστώ πάλι για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ και τους δύο για τις παρουσιάσεις σας, για τις απαντήσεις σας. Πολύ ενδιαφέρουσα και καρποφόρα ήταν αυτή η συζήτηση. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της Μαρχίας Διάταξης. Διορθωτικός προϋπολογισμός υπαρθμών 4 στο Γενικό Προϋπολογισμό του 2016. Επικαιροποίηση και τα λοιπά και τα λοιπά. Γνωρίζετε το ιστορικό. 11 Οκτωβρίου του 2016 οι συντονιστές συμφώνησαν ότι η Επιτροπή μας θα συντάξει γνωμοδότηση για το σχέδιο διευθυντικού προπολογισμού παρθυμών 4. Πρόκειται για μια από τι περιοδικέ επικαιροποίησει ε, του ετήσιου προπολογισμού τη Κομισιόν για να ληφθεί υπόψη εξελισσόμενο μοτίβο των ε, πληρωμών, αλήψεων υποχρεώσεων κτλ. Η Επιτροπή Προπολισμών Καθήλων Αρμόδια αποφάσισε να διαπραγματευτεί το σχέδιο διορθωτικού προπολισμού 4 με το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής για τον προπολισμό του 2017. Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια θα λάβει χώρα την 1η Δεκεμβρίου. Από αυτές τις συνθήκες η Επιτροπή μας δεν έχει επαρκή χρόνο για να συντάξει τελικά γνωμοδότηση. Επομένως, οι συντονιστές συμφώνησαν να συνταχθεί από μορφή επιστολή τη Προέδρου αυτή η γνωμοδότηση και να απευθυνθεί αυτή η επιστολή στον πρόεδρο τη Επιτροπή Προπολογισμών. Το σχέδιο ε, τη επιστολή το έχετε στα, στο φακελό σα. Συμφωνείτε με την προτινόμενη διαδικασία και με το σχέδιο επιστολή. Μ' ακούει και κανεί. Μ' ακούει ο κ. Να Ρόι. Ναι, είναι εξαιρετική επιστολή, λέει ο κ. Φανίστελ Ρόι. Thank you. really... Σας ευχαριστώ. Και πραγματικά εκπλήσωμαι που με ακούει έστω και ένας και που συμφωνεί και με την επιστολή μου. Ευχαριστώ. Κύριος Φανής Και ξαναπαίρνω πίσω τους δύο πόντους. Okay. Okay. Uh, so I close our... Άρα λίγη σημερινή συνεδρίαση και παρακαλώ να παραμείνουν οι συντονιστές με τη συνεδρίαση των συντονιστών να ακολουθείται κλεισμένο των θυρών. Οι μη έχοντες εργασία να αποχωρήσουν.